Okay, maybe we can take our seats, colleagues. Συνεχίζουμε συνάδελφοι, ξεκινάμε μάλλον για μια ακόμη φορά, πάντα με λίγη καθυστέρηση. Θα περάσουμε τώρα στο 12 προετοιμασία για τη συνάντηση ε, κορυφής για ανθρωπιστικά θέματα. Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 16 θα στείλουμε και αντιπροσωπεία. Τον Οκτώβριο ο μόνιμος εισηγητής θα μας παρουσιάσει μια έκθεση και θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα για 128 τροπολογίες και τις συμβιβαστικές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουερέρο λοιπόν για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι οι πολίτες του κόσμου, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφόρησης, συνειδητοποιούν ότι η ισόρευση ανθρωπιστικών κρίσεων στον κόσμο είναι ένα μήνυμα το οποίο δείχνει πώς είναι ο κόσμος μας σήμερα και σαν συνέπεια των κλιματολογικών αλλαγών δημιουργούνται κατεπίγουσες καταστάσεις, φυσικές καταστροφές ε, και υπάρχει και διάδοση βέβαια των συγκρούσεων και μη επίλυση ε, προβλημάτων τα οποία σωρεύονται και επηρεάζουν ε, τη ζωή των ανθρώπων όλο και περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουν όλοι οι πολίτες του κόσμου. Εμείς που αποτελούμε τμήμα αυτής της Επιτροπής ε, έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους για να συνειδητοποιήσουμε το βάρος αυτών των κρίσεων. Τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή αυτή καθοδηγούμενη από τον κύριο Γκέρεν ασχολήθηκε με, το, με την κρίση του έμπολα και εγώ και ο κύριος ε, Σέλα ασχοληθήκαμε με το θέμα της μείωσης ε, της προσπάθειας για μείωση των φυσικών καταστροφών η πρόεδρος ασχολήθηκε με τα θέματα της εκπαίδευσης, της ανθρωπιστικής κρίσης, όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε ε, και στα πλαίσια των στόχων του κυρίου Στίερ και στα πλαίσια της χρηματοδότησης του κυρίου Σίλβα Περέιρα και για τη συνάντηση κορυφής για το κλίμα της κυρίας Μακάβαν, όλα αυτά δείχνουν τη σχέση της στενή που έχουν με την ανθρωπιστική δράση και χαρακτηρίζουν συστηματικά τις εργασίες μας τους τελευταίους μήνες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, υπήρξε μια επαρκής πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή μας και υπήρξε μια στήριξη, θα έλεγα, για τα θέματα αυτά και στην Ολομέλεια. Και ακούστηκε έτσι η άποψη του Κοινοβουλίου γύρω από όλα αυτά τα προβλήματα και γύρω από όλες αυτές τις ε, δράσεις στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μπορέσει να εκφραστεί και σε σχέση με την ανθρωπιστική δράση και την ανθρωπιστική βοήθεια που θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη τον επόμενο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις απόψεις της με τη δική της ανασύνωση το Συμβούλιο στα τέλη του έτους, στις αρχές του επομένου θα εκφραστεί και αυτό και όλοι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια επιπλέον όθηση προς το Συμβούλιο και να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν συμμετέχουσα και διαπραγματεύτρια στη συνάντηση αυτή, συνάντηση κορυφής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του σεναρίου θέλω να ευχαριστήσω τους και όλους τις αλλά και όλους εσάς για τη συνεργασία σας, όχι μόνο τη συνεργασία αλλά την ενεργή συμμετοχή που είχατε όλοι γύρω από την έκθεση αυτή, γιατί το δεν αρκεί να παρουσιαστούν αυτές οι 125 τροπολογίες που εμπλουτίζουν το αρχικό κείμενο, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαπιστώνω ότι από τις 128 μάλλον αυτές οι 50 έχουν συνυπογραφεί από κοινού από τους σκιώδεις. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι σκιώδεις στην ουσία συνυπογράφουν την έκθεση αυτή και δεν είναι απλά σκιώδεις. Και υπάρχουν λοιπόν και 20 ε, συμβιβαστικές οι οποίες είναι καρπός της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Πάρα πολύ συχνά ε, νομίζω επεδείχθη η απαιτούμενη ευαισθησία δεκτικότητα από πλευράς των διαφόρων πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να αποφύγουμε οι μεν τις κόκκινες γραμμές των άλλων και να μείνουμε στα κοινά θέματα αυτά τα οποία μας ενώνουν. Συνέπεια αυτής της δραστηριότητας, συνέπεια της κατάθεσης αυτών των ε, τροπολογιών η έκθεση ενισχύει κάποια κομβικά θα έλεγα σημεία τα οποία γνωρίζουν πλέον καλά τα μέλη της Επιτροπής. Επιβεβαιούνται οι βασικές μας άρχες, ε, επίσης διασφαλίζεται ο σεβασμός των διεθνών κανόνων, εκφράζεται η σωστή αξιολόγηση των διεθνών ε, κανόνων ε, και καταδικάζεται η παραβίαση των κανόνων αυτών και αναφέρονται επίσης και τα προβλήματα και επιβεβαιώνονται λοιπόν και οι αρχές αλλά και γενικά το Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο. Τώρα για τη συγκεκριμένη προστασία των ομάδων εν κινδύνο, ε, δηλαδή γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι, ηλικιωμένοι. Βλέπουμε ότι οι δημογραφικά στοιχεία δείχνουν μια παράταση του προσδόκιμου ε, ζωής και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ειδικότερα προβλήματα των ανθρώπων αυτών και τα προβλήματα των εκτοπισμένων πληθυσμών αναγνωρίζεται ο, η σημασία και ο ρόλος των πληθυσμών που φύγονται από τις κρίσεις αυτές και όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα στα πλαίσια των κρίσεων αυτών, προσπαθούμε να δώσουμε μία απάντηση στα προβλήματα τα οποία τίθενται. Εκφράζεται και η επιθυμία να υπάρξουν επαρκή ανθρωπιστικά και οικονομικά μέσα για να υποστηριχθούν οι ΜΚΟ, οι τοπικές ΜΚΟ και για να υπάρξει μια θα έλεγα δυνατότητα πρόβλεψης για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων. Απαιτείται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να είναι πιο δραστήριες ε, και σε σχέση με τον έλεγχο των λογιστικών τους και να προετοιμάζουν με σωστό τρόπο και επαγγελματικό τρόπο ε, το προσωπικό τους. Στις χώρες δωρήτριες ε, ελπίζουμε να είναι να γίνει μια προσπάθεια ελάφρυνσης των γραφειοκρατικών βαρών που μας εμποδίζουν πολλές φορές να δώσουμε έγκαιρη απάντηση στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να είναι πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα, η ανιχνεσιμότητα και ο έλεγχος των λογαριασμών έτσι ώστε και των λογιστικών στοιχείων και σε σχέση με τη συνεργασία των κοινοτικών ταμείων με τοπικές αρχές και οργανώσεις με βάση την αρχή της αποτελεσματικότητας και την αρχή της συνεκτικότητας. Μαζί λοιπόν και με τις τροπολογίες και τις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν στις οκτώ συμβουλευτικές συναντήσεις οι οποίες προηγήθησαν για την προετοιμασία αυτής της συνάντησης κορυφής και τέλος θα ήθελα να πω ότι σε κάποια θέματα στα οποία υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες προσπαθήσαμε να βρούμε ένα επίπεδο συνεννόησης μέσα στο οποίο όλοι να μπορούν να ενταχθούν αποφεύγοντας οι αντίθετες θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων να προχωρήσουν σε μια παράλυση και να μπλοκάρουν την διαδικασία της έκθεσης αυτής. Γι' αυτό και συνεκλήθη μια συνάντηση με τους σκιώδεις προσπαθώντας να λύσουμε τα τελευταία προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε μέσω μιας συμβιβαστικής επιπλέον τροπολογίας. Θα ήθελα λοιπόν με κάθε ειλικρίνεια ε, να πω ότι εμείς παραμένουμε στοχευμένοι στην προσπάθειά μας και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε πάνω σε ένα θέμα στο οποίο είναι απαιτείται μάλλον να παρέμβουμε. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη από την βοήθειά μας να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους γιατί έτσι θα σεβαστούμε τους εαυτούς μας, τις ακίες, τις αξίες μας και τις αρχές μας. Ευχαριστώ. Θα δώσω πρώτο το λόγο στους της συζητητές. Ας ξεκινήσουμε τον κύριο Κέρενς. Έχω αρχικά τον Σάχλ, μετά την Χέιλι, μετά τον Ιγνάθιο, με αυτή τη σειρά. Σάχλ είχα νομίσει ότι ζητούσατε το λόγο. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε κάτι που για μας αποτελούσε κόκκινη γραμμή σε αυτή την έκθεση. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ιδίως σε εμπόλεμε ζώνες. Και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Θα πρέπει να δίνονται όλες οι, όλη απαραίτητη βοήθεια που χρειάζονται οι γυναικές, συμπεριλαμβανομένες και τη δυνατότητά τους να κάνουν έκτρωση όταν έχουν πέσει θύματα βιασμού. Εγώ γνωρίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι ευαίσθητο για πολλούς από τους συναδέλφους, αλλά ο Ερυθρό Σταυρός έχει υιοθετήσει αυτή την άποψη. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχει ε, εκφράσει και η κυρία Μογκερίνη. Γι' αυτό λοιπόν για εμάς αποτελεί κόκκινη γραμμή το θέμα αυτό και ήθελα να κάνω μια δεύτερη παρατήρηση πιο γενικού χαρακτήρα. Εδώ και ορισμένους μήνες παρακολουθούμε μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση να εξελίσσεται Ζητώ συγγνώμη που πάντα αναφέρομαι στο ζήτημα το χρηματοδότηση. Αλλά ήδη είχαμε μεγάλα προβλήματα με τη χρηματοδότηση εξαιτία του μεγάλου αριθμού των κρίσεων και των ε, πολεμικών συγκρούσεων. Αλλά πέρα από τους γνωστές συγκρούσεις τις οποίες ε, ε, συγκεντρώνει το φόντο της δημοσιότητας παραμένουν οι ε, κρίσεις οι ξεχασμένες στο Σουδάν, στην ε, Κεντρική Αφρική, στη Σάρα, στη, Μέση Ανατολή, πέρα από τη Συρία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται προς την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας είναι το εξής. Αυτή η κρίση προκαλεί προσφυγικές ροές που έχουν κόστος αντιμετώπισης στις χώρες υποδοχής. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση πολλές χώρες ανακοινώνουν ότι τα χρήματα τα οποία έδιναν για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια θα δεν θα τα δίνουν πια την αναπτυξιακή βοήθεια και θα τα χρησιμοποιήσουν για την υποδοχή των προσφύγων που έρχονται σε αυτές. Βεβαίως είναι μεγάλα τα έξοδα που δημιουργούνται για την υποδοχή των προσφύγων ε, στην, αμέσως μόλις έρχονται την πρώτη χρονιά, πράγματι. Αλλά με αυτή την ανακατονομή των πόρων θα βρεθούμε να μην έχουμε τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε άλλες κρίσεις. Το Ταμείο για τους καταβλισμούς στην Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει αποκτήσει ακόμα την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Πόσο γνωρίζω, και ενημερώστε με αν υπάρχουν και νέα στοιχεία, έφτανε μόνο το 1% την προηγούμενη εβδομάδα. η χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,8 δισεκατομμύρια πρόκειται για χρήματα τα οποία θα... Ε, δεν είναι νέα χρήματα, δεν είναι επιπλέον χρήματα, είναι χρήματα τα οποία θα αποκτηθούν από το Ταμείο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Το οποίο σημαίνει γενικά ότι το σύνολο των χρημάτων που είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των κρίσεων είναι περιορισμένο. η αντιμετώπιση που είδαμε στην Αντισάμπαμπα ε, κατά την άποψή μου δεν είναι αποδεκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει και μιλάει, ε, εκφράζει θέσεις οι οποίες ήταν, έχουν ήδη ξεπεραστεί. Πολλές χώρες είχαν ανακοινώσει μειώσεις της ε, χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή συνεργασία μέχρι και 40%. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε, εάν δεν σταματήσει αυτό, εάν δεν ε, βρεθούν επιπλέον πόροι, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ε, επαρκώς τις κρίσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλου τύπου ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως για παράδειγμα αντιμετώπιση της ελονοσίας ή της φυματίωσης σε ορισμένες ε, χώρες. Ε, πρέπει λοιπόν κατά την απόψή μου να σταματήσουμε αυτή την υποκρισία. Πρέπει να ζητήσουμε μια αύξηση των πόρων που δίνονται για την αναπτυξική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων κυρίως. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει το θέμα και να, να καταγγείλουμε το γεγονό ότι δεν υπάρχει απαιτούμενη πολιτική βούληση για να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το, βρίσκουμε και στην, το βλέπουμε και στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Εάν υπήρχε ε, ε, ε κατανομή των βαρών θα μπορούσαμε καλύτερα να την αντιμετωπίσουμε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον συνάδελφο Γερέρο ε, ότι θα αναδείξει αυτά τα ζητήματα, έχει την εμπειρία του μόνιμου εισηγητή. Έχει έρθει η στιγμή να ταρακουνήσουμε τους ηθήνοντες, δεν έχει νόημα να παριστάνουμε ότι υπάρχει συνένεση και ότι όλα βαίνουν καλώς. Όπως η υποτιθέμενη συνένεση που φαίνεται να υπάρχει από τις συναντήσεις των G7. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία ε, σε διάφορα φόρα τον επόμενο καιρό να θέσουμε τα ζητήματα αυτά. τη ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή και τους σκιώδη. Πιστεύω πως μπορούμε να συνεργαστούμε καλά. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως αναφέρθηκε σε αυτές και ο κύριος Γκέρεντς. Ο συμβιβασμός 14 αναφέρεται στην ερμηνεία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε περιπτώσεις όπου βιασμών ε, κοριτσιών και νέων γυναικών σε εμπόλεμες περιοχές. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δεν έχει να κάνει με το τι νομίζουμε εμείς. Έχει να κάνει με τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Οι γυναίκες και κορίτσια που είναι θύματα βιασμού σε εμπόλεμες χώρες υποφέρουν από πολύ σοβαρές συνέπειες αυτής της ε, πράξης και το να αρνούμαστε να τους ε, προσφέρουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και σε ασφαλείς ε, υπηρεσίες αμβλώσεων είναι κάτι απαράδεκτο. Πρέπει να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Και η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Επίτροπος Τηλιανίδης έχουν τοποθετηθεί από αυτού καθώς και αρκετοί ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει μια παρόμοια ερμηνεία του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Η συμβαστική πρόταση 14 λοιπόν θα έπρεπε, σύμφωνα με την δική μου πολιτική ομάδα, να μείνει όπως ε, συμφώνησαν οι σκιώδεις ηγητές στο Στρασβούργο. Και πιστεύω πως η δική μας Επιτροπή θα έπρεπε να τοποθετηθεί και να ζητήσει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα της μη συμμόρφωσης, της μη συμμόρφωσης από πάρα πολλούς φορείς αυτόν τον ε, καιρό σε πλαίσια διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Ιεμένη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν. Δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, ε, μια σοβαρή προειδοποίηση για την ε, συνεχόμενη παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και τώρα μάλιστα που συζητούμε για την ε, πρώτη διεθνή διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, πιστεύω θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τι γίνεται με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ, ο Ιγνάτσιο Κοράου. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκερέρο για την εξαιρετική του δουλειά με αυτή την έκθεση και για την εξαιρετική συνεργασία με όλους τους σκιώδες εισηγητές. Όπως ο Σαρλ Γκέρεντς και η Χέιντι Χάουταλα, οφείλω και εγώ να τονίσω αυτήν την κόκκινη γραμμή για τη συμβαστική πρόταση 14. Διότι όπως είπαν και εκείνοι, πρόκειται για διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν είναι κάποια προσωπική άποψη. Δεν μιλάμε για θρησκεία ή για άλλα θέματα που συνήθως ε, συζητούμε εδώ. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν μπορούμε να το συζητούμε έτσι με ελαφρότητα. Πέραν αυτών πρέπει να πω ότι θεωρώ την έκθεση πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα για τις δυνατότητες ε, που έχουμε να μεταφέρουμε αρμοδιότητες στα διεθνή ανθρωπιστικά φόρα, ιδιαίτερα τις δυνατότητες συντονισμού και φοδιαστικής που έχουμε. Εμείς υποβάλαμε 30 τροπολογίες, πολλές από αυτές με άλλους ασκιώδεις εισηγητές και εστιάζουμε περισσότερο στον αυτόχθονα πληθυσμό και σε άλλες ομάδες που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, ο Νταβοστίερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς, ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Θα... Τι να αντικαταστήσω, λοιπόν. Και θα ήθελα λοιπόν εκ μέρου του ΕΛΚ να ευχαριστήσω τον Ενρίκε για όλη την σκληρή δουλειά που έχει κάνει και τις προσπάθειές του να συμπεριλάβει όλες τις ε, διαφορετικές απόψεις που είχαμε. Υπήρξαν πολλές κόκκινες γραμμές από πολλούς. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν το έργο του. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι φιλοδοξία και του ΕΛΚ να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ψηφοφορίας τον οποίο να μπορέσουμε να εγκρίνουμε. Και να υπενθυμίσω ότι στις 12.30 θα έχουμε μια συνάντηση των σκιωδών όπου θα συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω και να σταθώ σε αυτά που είπε ο Σάρλ Γκέρενς και να ρωτήσω για την θέση του ΕΛΚ στι ε, διαπραγματεύσει. Μίλησα με πολλού εκπροσώπου μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Λέσβο και μου είπαν ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση με του ε, πρόσφυγε. και ο συντονισμός ε, δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού στις δικέ μα ανθρωπιστικέ προσπάθειε. Υπάρχουν πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που εργάζονται για αυτά τα θέματα και δεν μπορούν να συνεργαστούν σωστά. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ε, συζητήσει για αυτό το θέμα, αλλά όταν έχουμε ανθρωπιστικές κρίσεις στα ίδια μας τα εδάφη, αναρωτιέμαι πώς θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά θα έπρεπε να είναι η συντονίστρια αρχή, συντονιστική αρχή. και δραστηριοποιείται σε πολλά μέρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τι συμβαίνει και αν έχει κάποια πρόταση για έβρεση λύσεις. Ίσως ε, με τη βοήθεια κάποιων μεγάλων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον νότο της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ που θα μας ε, μιλήσει γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς στηρίζουμε το έργο που έχει ε, προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας για την έκθεση αυτή. Όπως είπε και ο κύριος Γερέρο, τώρα ε, συμπληρώνεται το παζλ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεκφράσει τη θέση της, το Συμβούλιο έχει προετοιμάσει συμπεράσματα, και τώρα έρχεται και το Κοινοβούλιο να εκφράσει τη θέση του για το ζητήματα αυτά. Για το ζήτημα που θίγεται, κυρία Πρόεδρε, για την εσωτερική, τον εσωτερικό συντονισμό, αναμένουμε ότι θα μας ασκήσουν κριτική ε, διάφορες συμμετέχοντες στη Σύνοδο της ε, Κωνσταντινούπολης και συζητούμε με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε εσωτερικά σε κρίσεις. Η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η λογική με την οποία προσέρχεται στη Σύνοδο είναι να δημιουργηθεί παγκοσμίω μια συμμαχία και ένα ένας για πρώτη φορά συζητούνται ε, στο επίπεδο των κρατών μελών τα ζητήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας στα ανθρωπιστικά και όλα τα κράτη-μέλη επιθυμούν να είναι επιτυχημένη η Σύνοδος. Θα προσπαθήσει να το ε, διευκολύνει αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνοντας το καλό παράδειγμα με την παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη. Κύριος Γερέρο. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και τους σκιώδεις εισηγητές και τον κύριο Στήρ που δεν είναι σκιώδης αλλά είναι σαν να ήταν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Σχετικά με την συνεδρίαση η οποία έχει συγκληθεί για τις 12.30 έχω την αίσθηση από τις διάφορες πολιτικές ομάδες ότι το περιθώριο κίνησης είναι πάρα πολύ μικρό και αν υπάρχει καν δηλαδή. Αλλά καλό είναι να δοκιμάσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε ικανοποιημένοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία, να ψηφίσουμε το απόγευμα για τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Γκέβεντς. Ο κύριος αναφέρθηκε σε μια γαλλική έκφραση, το coup de gueule, δηλαδή να ξυπνήσουμε μας περιπτώσει την προσοχή του άλλου. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και στα πλαίσια του ενεστώτος έτους που διαδέχονται η μία την άλλη διεθνείς συναντήσεις κορυφής αλλά δυστυχώς ε, τα θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση δεν τελειώνουν ποτέ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς, ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι κάθε φορά υψηλότερες. Ε, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία τέθηκαν ήδη και μπορούμε και εμείς συνολικά να θέσουμε. Το πρώτο, δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε οι νέες ανάγκες χρηματοδότησης να χρησιμοποιήσουν μέσα τα οποία ήδη έχει ορίσει, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλους τομείς. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη πιστώσεις οι οποίες ε, κανονικά θα έπρεπε να δοθούν σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς όπου χρειάζονται εξίσου. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τα ψηφίσματά μας μέχρι τη συνάντηση κορυφής της Κωνσταντινούπολης και η έκθεση που θα εγκρίνουμε στην Ολομέλεια τον μήνα Δεκέμβριο μέχρι όμως τον μήνα Μάιο με διαφορετικές πρωτοβουλίες, με προφορικές ερωτήσεις και με διαδοχικά ψηφίσματα να θέσουμε εκ νέου το θέμα της έκκλησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και προς το Συμβούλιο έτσι ώστε να προωθηθούν τα θέματα τα οποία θέτουμε εμείς και να συνεχίσουμε γενικά την προσπάθεια διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες. Και τρίτον, όπως είπε η Μακάβαν, Αύριο ξεκινά η συνάντηση κορυφή στην Βαλέτα, στη Μάλτα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Ε, ο τρόπος με τον οποίο εμείς βλέπουμε την Αφρική είναι περιορισμένος. Έχουμε από τη μία τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη Μέση Ανατολή, στη Μικρά Ασία μάλιστα λέει ο μιλητής, και σε συγκεκριμένες περιοχές της αραβικής σφαίρας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση στην Αφρική και ιδιαίτερα στην λεγόμενη υπόσαχαρική Αφρική περιλαμβάνει πολεμικές συγκρούσεις, περιλαμβάνει αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ίσως εξίσου σημαντικό και επηρεάζει με τρόπο εξίσου σημαντικό ε, τα προβλήματα που δημιουργούν ε, οι ανθρωπιστικές αυτές κρίσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και δεν φτάνει να μετακινούμε κάποιες πιστώσεις από προηγούμενες δράσεις σε καινούργιες. Θα στηρίξω λοιπόν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκέρενς και τις πρωτοβουλίες μας τις οποίες θα πρέπει να συνεχίσουμε, ό,τι πρωτοβουλίες είναι αυτές έτσι ώστε να επιστήσουμε την προσοχή των εμπλεκομένων στα προβλήματα αυτά. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει ένα υψηλότατο βαθμό σύγχυσης. Η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων εκτός των συνόρων μας, ενώ τώρα Προσπαθούμε, καλός ή κακός, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και τα ανθρωπιστικά προβλήματα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσουν με ευθύνη και δύναμη πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Το τελευταίο θέμα είναι η προετοιμασία για τη συνάντηση κορυφής για το κλίμα και η χρηματοδότηση των υποανάπτυξη χωρών σε σχέση με τέτοιου είδους θέματα που συνδέονται με το κλίμα, τίθενται θέματα προσθετικότητας, τίθεται το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τα προβλήματα αυτά, θα τα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και για τα θέματα της ασφάλειας στην Αφρική τον μήνα Δεκέμβριο διοργανώνουμε μία ακρόαση για το κέρας της Αφρικής πιο συγκεκριμένα. Από ό,τι φαίνεται στο βορρά της Αιθιοπίας υπάρχει πλέον λιμός και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε, ίσως θα πρέπει να φτάσουν στην Ολομέλεια και να δούμε συνολικότερα το πρόβλημα γενικά της μετανάστευσης. Εν πάση περιπτώσει θα ψηφιστεί το απόγευμα η έκθεση αυτή και θυμίζω και την συγκεκριμένη συνάντηση στις 12.30. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα είναι σύντομο νομίζω, είναι το 13 έκθεση για που την οποία κάναμε στο Μιλάνο για την Expo Μιλάνο ενέργεια για τη ζωή και η κυρία Ζαμπόσκα και άλλοι συνάδελφοι ήταν παρόντες ε, ξέρετε ότι κάθε δύο χρόνια διοργανώνεται ένα τέτοιο συμβάν. Η Επιτροπή μας προσεκλήθη λόγω του θέματος το οποίο είχε επιλεγεί φέτος στην παγκόσμια αυτή έκθεση. Τροφοδοσία του πλανήτη, τρόφιμα για τον πλανήτη, ενέργεια για τη ζωή. Τέθηκε το θέμα της ε, ασφάλειας ε, στον τομέα της προμήθειας τροφίμων, τέθηκε το θέμα της επιστικής βοήθειας, ο Μπανκιμούν έκανε μια τεράστια συνάντηση, οργάνωσε μια τεράστια συνάντηση υψηλού επίπεδου με πάρα πολλούς εκπροσώπους, αρχηγούς κρατών. Εμείς οργανώσαμε κάποιες συναντήσεις επιμέρους για θέματα δικαιωμάτων των πληθυσμών, επίσης θέματα ιδιοκτησίας γης, Έχουμε τον Σενάν Γκουσμάου μαζί μας, τον πρώτο πρόεδρο του Ανατολικού Τιμόρ ε, και τον είχαμε εκεί και παρουσίασε τη χώρα του, βοήθησε στη χώρα του να δημιουργηθούν δημοκρατικές δομές μετά από τον δύσκολο αγώνα εναντίον της κατοχής της Ινδονησίας. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος αλλά και διασκεδαστικός άνθρωπος είναι σίγουρα κάποιος ο οποίος αξίζει ιδιαίτερη αναγνώριση. Συζητήσαμε τα πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, όπως σαν παράδειγμα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, Τέθηκαν ερωτήσεις προς τον κύριο Γκουσμάο για το αν σαν παράδειγμα θα πρέπει να υπάρξουν μετακινήσεις πληθυσμών για να εκμεταλλευτούμε εμπορικά τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ε, και τέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους φοιτητές μάλλον του Πανεπιστημίου της Βενετίας. Είχαμε ε, την κυρία Τέγκεν που είναι μια μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση ε, έχεις μέσω της οποίας επιβιώνει στην Αιθιοπία. Ε, είπε ότι οι γυναίκες συντηρούν αυτές τις μονάδες και οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες διασφαλίζουν την επιβίωση της οικογένειας. επισκεφθήκαμε και τα περίπτερα διαφόρων χωρών και αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον είναι ότι έθεταν το θέμα της αηφορίας και των στόχων της χιλιετίας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμείς να βλέπουμε το πόσο αλληλένδετα είναι όλα αυτά τα συστήματα. Ιταλικό περίπτερο, γαλλικό, βρετανικό και άλλες χώρες ήταν μια καλή αποστολή θα έλεγα. Η γραμματεία την οργάνωσε πάρα πολύ καλά και είναι νομίζω ένα σωστό θεμέλιο για την έκθεση που θα κάνουμε εμείς για την διασφάλιση προμήθειας τροφίμων για την Αφρική και για τους λοιμούς που μαστίζουν την Αφρική θα μας βοηθήσει η επίσκεψη αυτή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η Χάιντι νομίζω ότι μας παρουσίασες με καλό τρόπο τα θέματα της συμμετοχής της Επιτροπής μας. για τα δικαιώματα στη γη. Ε, τα πάνελ είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη και ίσως στα πλαίσια των διαφόρων προτεραιοτήτων μας μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Βέβαια η έκθεση Χόιμπουκ για την ασφάλεια στην προμήθεια τροφίμων είναι το κεντρικό σημείο, αλλά παρόλα αυτά ίσως να υπάρχει δυνατότητα να το συζητήσουμε και αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ολοκληρωμένη η παρουσίαση που μας έκανες. Ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να αναφέρω. Τα τρόφιμα για τον πλανήτη πρέπει να συνδέονται με το πόσιμο νερό και αυτό προτείνω να αναφέρουμε από εδώ και στο εξή σε όλες τις εκθέσεις ή τις γνωμοδοτήσεις που θα συντάσσουμε στο Κοινοβούλιο. Κάποιες χώρες, ξέρετε, θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα, μεγάλες ελλείψεις νερού όχι μόνο πόσιμου νερού, αλλά και νερού για την παραγωγή τροφίμων. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί απασχολεί όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα το συνδέσουμε αυτό και με το θέμα απόψε το απόγευμα για την κλιματική αλλαγή και τα τρόφιμα. Θα αναφερθούμε στην ξηρασία, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα, συνεχίζουν και εξακολουθούν να εμφανίζονται και πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε για να βρούμε μια βιώσιμη λύση. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Όχι, ο κύριος ε, Σακέο φαίνεται πως δεν είναι εδώ. Πολύ ωραία συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε την έκθεση Χόιμπουχ και θα συζητήσουμε με τους συντονιστές για το θέμα των δικαιωμάτων στη γη και στο νερό. Περνάμε τώρα στο σημείο 14, εφαρμογή της ε, στρατηγικής για την ε, Κεντρική Ασία. Είναι μια γνωμοδότηση ε, έκθεση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριο Σόπφλιν είναι ο εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως η έκθεση είναι αρκετά καλή. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Ε, να πω το εξής. Έχω την εντύπωση πως δεν είναι έτοιμες όλες οι μεταφράσεις της γνωμοδότησης. Υπάρχει αγγλική εκδοχή, διότι στα αγγλικά την έγραψα την γνωμοδότηση, όμως νομίζω πως δεν έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε για να έχουν πρόσβαση όλοι. Ξέρετε, δεν μιλούν όλοι αγγλικά. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, λογικά οι μεταφράσει θα πρέπει να είναι έτοιμες αυτή την εβδομάδα, αλλά με το που τελειώσετε την παρουσίαση θα ξέρω περισσότερα. Πιστεύω πως ε, η Κεντρική Ασία, δηλαδή το Τούρκισταν και οι υπόλοιπες χώρε ε, στάν της περιοχής, είναι ε, περιοχή με πρώην απικίες και η δομή ε, των ε, χωρών αυτών ήταν έτσι ώστε να ωφελήσουν τη Σοβιετική Ένωση και όχι τις ίδιες τις ε, χώρες. Μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι απομακρυσμένες, απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από οποιοδήποτε μεγάλο κέντρο. Για να πάτε ας πούμε από τη Μόσχα στο Καζακστάν η πτήση διαρκεί 4 ώρες φανταστείτε. Και το 1991 λοιπόν ήταν αναμενόμενο αυτές οι χώρες να ανεξαρτητοποιηθούν, κάτι που δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν ήταν έτοιμες να ε, αναλάβουν τις ε, πλήρες αρμοδιότητες που απαιτεί ένα ανεξάρτητο κράτος. Επίσης, ο πληθυσμός των ε, χωρών αυτών, ιδιαίτερα του Καζακστάν, αποτελείται από επίκους. Για παράδειγμα, το 40% των κατοίκων του Καζακστάν είναι Ρώσοι. και υπάρχουν πάρα πολλοί στην ε, Ρωσία που πιστεύουν ότι το Καζακστάν είναι μια σλαβική χώρα και θα πρέπει να προσαρτηθεί ξανά στη Ρωσία. Έπειτα ένα θέμα ακόμα είναι και η οικονομική ανεξαρτησία. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Καζακστάν το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ε, σοβαρό. αλλά όχι μόνο στο Καζακστάν. Το 50% των εσόδων της οικονομίας του ε, Τατζικιστάν προερχόταν από την ε, Ρωσία. Αλλά νομίζω πως ε, και κάποιες άλλες χώρες της περιοχής είναι σε παρόμοια κατάσταση. Κυργυσία, για παράδειγμα. Ε, επίσης μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία αλλά και όχι μόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα στην περιοχή, ιδιαίτερα στις γειτονικέ ε, με το Αφγανιστάν χώρες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μεγάλες δυνάμεις οι οποίες παίζουν διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια. Η Κίνα επίσης ενδιαφέρεται για την περιοχή, όχι τόσο για λόγους στρατηγικής αλλά για πρώτες ύλες από τις χώρες αυτές. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως ε, υπήρχε διαμάχη ανάμεσα στην τσαρική Ρωσία και την εκείνα το 18ο και 19ο αιώνα και αυτές οι εντάσεις επικρατούν κατά πολύ και σήμερα. Υπάρχουν διάφορες ε, περιοχές οι οποίες επίσης έχουν έφορα εδάφη και ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ρωσία. Επίσης, οι γλώσσες που ομιλούνται στην περιοχή δεν έχουν ξεκάθαρα όρια, οπότε περιπλέκονται τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Και μην ξεχνάμε πως δεν υπάρχει κάποιος επίσημος μηχανισμός επίλυσης ε, κρίσεων στην περιοχή, κάτι που ωφελεί τη Ρωσία περισσότερο από όλους. Η Ρωσία λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο Τώρα, ας πάμε στην περίπτωση του Ουσμπεκιστάν. Το Ουσμπεκιστάν είναι η μεγαλύτερη χώρα από τις ε, υπόλοιπες της περιοχής και αναμένει να έχει ηγετικό ρόλο. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόβλημα, διότι αν ε, δούμε τον χάρτη και τον συγκρίνουμε με τους ε, χάρτες της περιοχής από 100-150 χρόνια πριν, θα δούμε ότι έχουν συρρυκνωθεί οι χώρες αυτές. Επίσης, ας μην ξεχνάμε τις παραβιάσεις ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων που έχουν λάβει χώρα από τη Σοβιετική Ένωση. Και ως ε, εμπειρογνώμων για την ε, περιοχή αυτή θα ήθελα να πω πως πρόκειται για πάρα πολύ σεισμογενής περιοχής και πρέπει να περιμένουμε κάποιες μεγάλες καταστροφές. Στην Τασκένδη, για παράδειγμα, είχε συμβεί πριν ένας μεγάλος σεισμός πριν από μερικές δεκαετίες με καταστροφικά αποτελέσματα. Τώρα, εγώ θα πρότεινα να γίνει μια γενικότερη μεταστροφή προς το κράτος δικαίου. Ο εκδημοκρατισμός των χωρών αυτών επίσης καθυστερεί αρκετά. Και ας μην ξεχνάμε ότι και οι κοινωνικές δομές είναι τελείως διαφορετικές. Είναι κυρίως οικογενειοκρατική κοινωνία αυτή των χωρών αυτών και Ξέρω ότι για παράδειγμα, στο Καζακστάν, εξαιτία ε, ε, των μεγάλων ε, βαθμών συγγένειας, απαγορεύονται οι γάμοι ανάμεσα σε συγγενείς μέχρι 7 βαθμούς συγγένειας. Κάτι άλλο επίσης που είναι πολύ δύσκολο και πολύ διαφορετικό από τις συνήθες πρακτικές που γνωρίζουμε είναι το ζήτημα της ηθαγένειας στις χώρες αυτές. Έχουν πολύ διαφορετικά έθιμα από εμάς και επίσης η διαφθορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρετε, η οικογένεια έχει ε, περισσότερη βαρύτητα από την αξιοκρατία στις χώρες αυτές και αυτό επίσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως και έχει δημιουργήσει. Μεταξύ άλλων προβλήματα εθνικής πόλωσης. Τώρα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει κάποια βοήθεια στην περιοχή αυτή, κυρίως οικονομική, όμως από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα μοτίβο ε, άσχημο, παιδική εργασία. Στέλνουν τα παιδιά να δουλέψουν ε, στα χωράφια, να βοηθήσουν στη συγκομιδή βαμβακιού. Δεν έχουμε διαπιστώσει αν αληθεύουν τα στοιχεία που έχουμε, όμως ε, αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Επίσης, αυτά είναι λίγα μόνο από τα ευρήματά μου στην Κεντρική Ασία και για περισσότερες πληροφορίες ε, με τα χαράς να σας ε, μιλήσω παραπάνω. Ο κύριος Τσέλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. έχει επικεντρωθεί στο παρελθόν και στο παρόν των χωρών αυτών της Κεντρικής Ασίας. Ωστόσο πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω πως μου λείπει η αναφορά στην αναπτυξιακή πολιτική, δηλαδή η άμεση σχέση της δικής μας Επιτροπής, της Επιτροπής Ανάπτυξης και πιστεύω πως ε, πρέπει να συμπεριληφθεί, διότι η περιοχή της Κεντρικής ε, Ασία ε, για μας δεν είναι κάτι αδιάφορο, είναι μια πολύ σημαντική γεωπολιτικά περιοχή. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και το Αφγανιστάν και ε, ωστόσο διαφέρει πάρα πολύ από όλες αυτές τις χώρες. Πέρυσι πήγαμε μια αντιπροσωπεία της ε, Κεντρικής Ασίας στο Καζακστάν, στο Τατζικιστάν και στην Κυργυσία. Παρακολουθήσαμε την εκλογική διαδικασία εκεί και είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ακόμα και ανάμεσα σε αυτές τις χώρε. Η Κυργησία για παράδειγμα, έχει ένα πολυκομματικό ε, σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα κράτη όχι. Τα υπόλοιπα κράτη διοικούνται από προέδρους που, για να το πω έτσι απαλά, είναι απολυταρχικοί. Επίσης, Υπάρχουν διαφορετικές ε, οικονομίες στις χώρες αυτές ε, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το Καζακστάν, για παράδειγμα, και το Τουρκμενιστάν δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην ε, αναπτυξιακή μας πολιτική, διότι το Καζακστάν έχει ένα οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο πλέον, το οποίο το κατατάσσει στην ανώτερη μεσαία τάξη των αναπτυξιακών προτύπων. Το Τουρκμενιστάν είναι ένα λίγο πολύ απομονωμένο κράτος, το οποίο έχει φυσικά μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όμως ο πληθυσμός δεν απολαμβάνει την ίδια ποιότητα ζωής με άλλα αντίστοιχα πλούσια σε φυσικούς πόρους κράτη. Στηρίζω βέβαια το να δίνουμε οικονομική βοήθεια σε τέτοια κράτη, όμως ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν αυτές οι διαφορέ Τώρα, τα Ουσμπεκιστάν, αυτές οι χώρες εμαστίζονται από φτώχεια. Πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες για την καταπολέμηση της και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Σόπφλιν επίση μα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση στο Ουσμπεκιστάν. Υπάρχουν ε, το 35% μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, του ΑΕΠ του, της χώρας αυτής προέρχεται από συνάλλαγμα, από μετανάστες που στέλνουν το προϊόντα της εργασίας τους από το εξωτερικό. Και επίσης υπάρχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, υπάρχει πρόβλημα με ναρκωτικά στην χώρα αυτή και καταλαβαίνετε πως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές αυτές τις χώρες. Η χρηματοδότηση λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να επαναξετάσουμε, καθώς και οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν πως πρέπει να συζητήσουμε το πού πηγαίνουν τα χρήματα και να μην ξεχνάμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να πηγαίνει στους πολίτες όχι στις κυβερνήσεις τους. Μην ξεχνάτε πόσο απολυταρχικές είναι και αυτές οι κυβερνήσεις και ο κύριος Σόπφλιν το είπε εξάλλου, οι χώρες αυτές μαστίζονται από διαφθορά σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Και δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς και οι κάτοικοι των ε, χωρών αυτών. Είναι λοιπόν ε, πολύ σοβαρή η πολιτική διάσταση του θέματος και πρέπει να ληφθεί εξίσου σοβαρά υπόψη στην γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόιζερ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους του Άρνε Λίτς, ο οποίος δεν μπόρεσε δυστυχώς να έρθει σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Και θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Τσέλερ και να πω ότι έχουμε μία περιοχή η οποία έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές ε, κατά τη διάρκεια των ε, χρόνων, των αιώνων. Πριν από 25 χρόνια, οι χώρες αυτές απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από τη Σοβιετική Ένωση. Πολλές δεν ήταν έτοιμες για να την αποκτήσουν. Βλέπουμε τώρα ότι μόνο δύο από αυτές, το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν δηλαδή, έχουν προχωρήσει έχουν προοδεύσει, έχουν φτάσει σε καλό σημείο. Οι άλλες όμως τρεις χώρες, η Κυργυσία, το Τατζικιστάν και το Ουσπεκιστάν, απέχουν πάρα πολύ από τα υψηλά επίπεδα ζωής των, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν μάλλον και του Καζακστάν. Χρειάζεται λοιπόν να καταβληθούν μεγάλε προσπάθειε και στην κοινωνία των πολιτών και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δική μα οικονομική βοήθεια. Πρέπει να σταθούμε επίσης σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, ε, να σταθούμε στην γεωργία, στις χώρες αυτές και στο πρόβλημα της ε, ίδρευσης. Διότι το πρόβλημα του νερού και της ελλειψητρίας θα μπορούσε να εντείνει τα προβλήματα των χωρών αυτών. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες για καλύτερη συνεργασία και επίσης να συμπεριληφθούν και οι γειτονικέ μεγάλες δυνάμεις και η Ρωσία και η Κίνα στο, στην προσπάθεια αυτή. Ας μην ξεχνάμε πως όπως είπατε και οι προηγούμενοι υπάρχουν πολλά συμφέροντα στην περιοχή αυτή, ιδιαίτερα επειδή γειτονεύουν με το Αφγανιστάν. Ας σταθούμε λοιπόν σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική με ιδιαίτερη εστίαση στο θέμα του νερού και των θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα το πρόβλημα του νερού, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αιτία σειράξεων στο μέλλον. Υπάρχουν διάφορες ε, αναταραχές επίσης στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα στις χώρες ε, οι οποίες εξαρτώνται απόλυτα από το ξενοσυνάλλαγμα των ε, μεταναστών τους που εργάζονται στη Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη πιθανά η κατάσταση αυτή λοιπόν στις χώρες αυτές. Και πρέπει να το έχουμε αυτό σοβαρά υπόψη μας ε, στην χάραξη της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Η εισαγωγή στη γνωμοδότηση που έχει συγγράψει ο εισηγητής δείχνει την βαθιά γνώση του για την ιστορία αυτής της περιοχής. Εμείς προτείνουμε λίγες τροπολογίες παρόμοια για να ε, δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ανέφεραν στην, ε, στην αναπτυξιακή συνεργασία και σε όλα αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει για αυτήν την περιοχή αλλά τα σημαντικότερα ήδη αναφέρονται στο προσχέδιο εκθέσης του κυρίου Σουέπφλιν. Εγώ θα ήθελα απλώ να τονίσω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για μια βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το Τατζικιστάν και το, Κυριστάν έχουν φτάσει στα πρόθυρα του πολέμου εξαιτία της... του χειρισμού των... Ε, ε, του νερού μεταξύ τους. Και φυσικά η κλιματική αλλαγή είναι ένα ε, ζήτημα πολύ σημαντικό εδώ όταν έχουμε βουνά στο Τατζικιστάν 6.000 μέτρων σιγά σιγά να λιώνουν τα χιόνια ε, στις κορυφές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής πρέπει να περιμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια η σύγκρουση για το νερό θα γίνει ακόμα εντονότερη και θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, των αρχών σε αυτές τις χώρες, για τη σημασία της διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων, ε, για να μην βρεθούμε σε καταστάσεις ε, όπου η σύγκρουση για το νερό να οδηγήσει μέχρι και σε πολέμους. Αναφέρθηκε ήδη ότι ε, πολλές από αυτές τις χώρες εξαρτώνται από την εισρωή συναλλάγματος από τους μετανάστες και αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις και στις κοινωνικές δομές. Η Φινλανδία έχει υποστηρίξει την, ε, τα δίκαια αιτήματα των ε, γυναικών ε, που έχουν μείνει πίσω ενώ οι άντρες τους έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και... Γιατί συχνά, εάν δεν είχαν ε, ε, δεν ήταν ε, παντρεμένες με τους ε, σύζυγους τους, ε, βρίσκονται χωρίς καμία κοινωνική προστασία. Και βεβαίω οι κακέ σχέσει αυτών των χωρών με τη Ρωσία είναι ε, ακόμα ένα παράγοντα που έχουν συμβάλει στην, ε, στην μη σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων και στην ανεργία στην περιοχή. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την άνοδο του βίου εξτρεμισμού που διαπιστώνουμε να συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές και το ονομαζόμενο Ισλαμικό κράτος προσπαθεί να επεκτείνει τα πλοκάμια του σε αυτές τις περιοχές στην Κεντρική Ασία. συνεχίζεται η βοήθεια η τομεακή, η οικονομική προς το Κυριστάν και το Τουρκμενικιστάν. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτή η χρηματοδότηση να συνδεθεί περισσότερο με το αίτημά μας να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις και κυρίως καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίση θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν αναλυφθεί σημαντικές πρωτοβουλίε για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ε, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία η λεγόμενη EIT που προσπαθεί να, δώσει, να, υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο οι, οι εξορρυκτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς. αναφέρθηκε το ζήτημα της ξαναγκαστικής εργασίας. Ιδίως όσον αφορά το Ουσμπεκιστάν, αυτό είναι ένα ζήτημα χρόνιο και οι αρχές του Ουσμπεκιστάν, η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν δεν μας έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις ε, για το πώς καταπολεμά και πώς ε, θα σταματήσει την ε, ξαναγκαστική εργασία παιδιών στα, ε, στις βαβακιού. Αυτά κυρίε σημεία από μένα. Βεβαίω το συνεργαστώ με τον εισηγητή για τα ζητήματα που ανέφερα. Κυρία Βαρίνα. Κυρίω Βαρίνα. Το προσχέδιο της έκθεσης του κ. Σέφιλτ είναι καλή βάση για να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση. Εγώ θα ήθελα να τονίσουμε περισσότερο τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας σε αυτή τη γνωμοδότηση. Εγώ έχω προτείνει τρεις ε, τροπολογίες. Η πρώτη αναφέρει ότι υπάρχουν παραδοσιακά συνεργασίες μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας και αυτές οι συνεργασίες, αυτό το δίκτυο συνεργασιών θα έπρεπε να, ενισχυθεί. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών είναι για εμένα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Δεύτερον, ε, ζητώ να υπάρξει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρωτοβουλειών των κρατών μελών ε, Γνωρίζω και με την προηγούμενη με οδιότητα του Υπουργού για την Αναπτυξιακή Συνεργασία στη Φινλανδία. Είχαμε ξεκινήσει ένα ε, πρόγραμμα ε, βοήθειας προς τις, ε, τα νέα ανεξάρτητα κράτη που είχαν προκύψει μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και άλλα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των κρατών μέλων που αναλαμβάνονται τις πρωτοβουλίες. Και βεβαίω υπάρχει και η συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τις ΗΠΑ, την οποία θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε και στην περιοχή. Και η τρίτη τροπολογία ε, προτείνει να προσθέσουμε μια αναφορά στην ε, συνεργασία με τα ταμεία τα αναπτυξιακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της, την Παγκόσμια Τράπεζα. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε ακριβώς στην αγνόηση της ε, διαφοροποίησης αυτής. Ο κύριος Ζέλερ αναφέρθηκε στο πρόβλημα θυμίζοντας ότι κάποιες χώρες δεν παίρνουν πλέον βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας την οποία έχουμε στηρίξει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου είναι το να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της ε, εφαρμογής της αρχής επικουρικότητας. Κάποιες ασθένειες όπως ε, η, ε, η φυματίωση συνεχίζουν ε, να καλπάζουν σε κάποιες χώρες της λεγόμενης της τέος Σοβιετικής Ένωσης και έχει υπάρξει και το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά είναι κάτι το οποίο απειλεί τους πληθυσμούς των χωρών αυτών αλλά φυσικά απειλεί και εμάς τους ίδιους. Η αρχή της επικουρικότητας όμως δεν μας επιτρέπει να παρέμβουμε. Το Ταμείο Καταπολέμησης του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας αναφέρεται σε αυτό λέγοντας ότι η φροντίδα η οποία δίδεται στις χώρες αυτές θα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της στρατηγικής μας εμείς. Νομίζω ότι το θέμα της υγείας είναι θέμα κοινού συμφέροντος και διαρωτώ με αν ο εισηγητής μετά και από τη διαφώτιση πιθανώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δεχθεί μια τροπολογία γύρω από αυτό. Ξέρω ότι οι διεθνείς οργανώσεις θα ήθελαν να παρέμβουν αλλά δεν μπορούν να το κάνουν πλέον λόγω ακριβώς ε, επαρκούς τροφοδοσίας οικονομικής για τα θέματα στα οποία προαναφέρθηκα. Ο Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι στην ώρα μου γιατί έπρεπε να είμαι σκιώδης εισηγητής και κάπου αλλού. Λοιπόν, έχω και εγώ κάποια πράγματα να πω, να προσθέσω μάλλον στις ε, απόψεις που ακούστηκαν ήδη ε, και να πω ότι πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πιο συγκεκριμένοι δηλαδή αναφερόμενοι στα προβλήματα της Κεντρικής Ασίας. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης πιστεύω πως είναι πολύ γενικό, δηλαδή μας κάνει μια ιστορική αναδρομή, μας παρουσιάζει τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή ανά τους αιώνες. Εντάξει, είναι βέβαια σχετικό και χρήσιμο, όμως όχι για την μελλοντική χάραξη της πολιτικής μας στην Κεντρική Ασία και πιστεύω επομένως πως η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να σταθεί στις οικονομικές εξελίξεις, στις αγορές πρώτων υλών συγκεκριμένα. Διότι ας μην ξεχνάμε πως εδώ πρόκειται για χώρες οι οποίες ε, ε, για πάρα πολλά χρόνια εποφελήθηκαν από τις αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών και τώρα από το 2013 δηλαδή και έπειτα η κατάσταση αυτή ε, έχει αλλάξει, έχουν, ε, έχει επιδεινωθεί η οικονομική τους ε, κατάσταση λόγω των αλλαγών στην αγορά πρώτων υλών και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλη αποδυνάμωση της οικονομικής τους δραστηριότητας, κυρίως εξαιτία των οικονομικών δραστηριοτήτων της ε, Κίνας που έχει δημιουργήσει μικρότερη ζήτηση σε πρώτες Και πρέπει να κατονομαστεί πιστεύω αυτό το πρόβλημα στην γνωμοδότησή μας. Επιπλέον, πρέπει να γίνει μια διαπίστωση ότι παρά δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης επιμένει το πρόβλημα της φτώχειας, ε, το οποίο είναι μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο σε αυτές τις χώρες. Το πρόβλημα αυτό οδηγεί σε τεράστιες εισοδηματικές ανισότητες αλλά και από την άποψη της υγείας. Ήδη ο κύριος Γκέρενς μας είπε πως υπάρχει μικρό προσδόκιμο ζωής, ιδιαίτερα για τις ε, πιο φτωχές περιοχές, για την Ήπεθρο, για τις ε, πιο ευάλωτες ε, πληθυσμιακές ομάδες και πιστεύω πως ε, πρέπει η αναπτυξιακή μας πολιτική να έχει αυτό ως ε, γνώμονα, ως κεντρικό σημείο. Τις ε, περιοχές δηλαδή που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, τις περιοχές που μαστίζονται από την φυγή των πολιτών. Οι άντρες πηγαίνουν προς τα αστικά κέντρα, μεταναστεύουν, οι γυναίκες μένουν πίσω και δεν μπορούν να έχουν ένα, μια καλή ποιότητα ζωής. Έπειτα, ένα στοιχείο που πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αναπτυξιακή αλλά και την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μεγαλύτερη ένταξη περιφερειών της Κεντρικής ε, Ασίας. Η μεγαλύτερη τους ένταξη και σε υποδομές ε, και στον χώρο των μεταφορών. Πρέπει να βελτιωθούν δηλαδή οι υποδομές και στις μεταφορές έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση σε ορισμένες από αυτές τις ε, περιφέρειες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί έμφαση στις ε, υπηρεσίες μεταφορών, στις υπηρεσίες υποδομών, στην ε, ενίσχυση των ε, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους ε, τομείς, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δικτύωση των περιφερειών αυτών. Αυτά προς το παρόν ε, από εμένα για τις παρατηρήσεις μου και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσέλερ θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Ναι, να συνεχίσω αυτό που είπε ο κύριος ε, Γκέρεν. Στο Κυργιστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κυργιστάν χρειάζονται βοήθεια και στην ε, διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και στην ε, γεωργία. Αλλά και στο θέμα της υγείας, της, της φαρμακευτικής περίθαλψης. Υπάρχουν μεγάλες απειλές για αυτές τις χώρες από έλλειψη υδάτινων πόρων, από έλλειψη τροφίμων, από έλλειψη σωστής υγειονομικής περίθαλψης και να μην ξεχάσουμε επίσης και την ε, κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό έχει ως συνέπεια μεγάλα προβλήματα υγείας, έχει συνέπεια ασθένειες, τη φυματίωση για παράδειγμα που αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο. Χρειάζεται επίσης να δοθεί έμφαση στην μεγάλη διαφθορά, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας αυτές τις χώρες και χρειάζεται μεγάλη προσοχή τα η οικονομική βοήθεια να πηγαίνει πραγματικά στους ε, δικαιούχους της, στους πολίτες. Επίσης πρέπει να ασκήσουμε κριτική και στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Ας μην ξεχνάμε βέβαια πως αυτές οι κυβερνήσεις έχουν διαφορετικές σχέσεις με τις ε, μεγάλες δυνάμεις, με την Ρωσία για παράδειγμα. Υπάρχει μια τελωνιακή ένωση με την ε, Ρωσία. και μάλιστα βρίσκονται λίγο πριν την ε, υπογραφή συμφώνου περισσότερης ε, ένωσης με τη Ρωσία, το Καζακστάν για παράδειγμα. Και να επαναλάβω τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν ε, είναι πιο ανεπτυγμένες από τις άλλες τρεις. Και όσον αφορά τους ε, μετανάστες, 5 εκατομμύρια μετανάστες εργάζονται στη Ρωσία από αυτές τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και χωρίς το συνάλλαγμά τους θα καταρρεύσουν οικονομικά οι χώρες αυτές. Και αν καταρρεύσουν οικονομικά τότε θα χτυπήσουν άλλες πόρτες και να αναφερθώ και στο πρόβλημα του Ισλαμικού κράτους. Ξέρετε, βρίσκεται πρώτον πυλών. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διεισδύσουν στην Κεντρική Ασία. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες Κεντρικής Ασίας είναι μουσουλμανικές χώρες. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα και να τα προσθέσουμε στα ήδη υπάρχοντα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτό δεν ξεφεύγει της προσοχής των Πολιτειών. Μην ξεχνάτε κιόλας ότι ο, και, ο αντιπρόεδρος Κέρι πέρασε μια ολόκληρη μέρα στο Τατζικιστάν συζητώντας αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Και όντως ε, καλά που αναφερθήκατε στο πρόβλημα του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχει κάποιος ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, εδώ είστε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα με την Κεντρική Ασία. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την αλλαγή αυτή από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ πρώτα. Πράγματι η Κεντρική Ασία θεωρείται περιοχή μεγάλης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα βασικό συστατικό είναι η αρχή της διαφοροποίησης, γιατί είναι διαφορετικές οι πέντε αυτές χώρες μεταξύ τους. Θέλουν να διακριθούν, να ξεχωρίσουν από τους γείτονές τους, έχουν διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας και θέλουν όλες να προχωρήσουν τις διμερείς μας σχέσεις. Έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις μας λοιπόν μία όθηση η οποία θα μας βοηθήσει να ορίσουμε καλύτερα και να τονώσουμε τις μορφές συνεργασίας μαζί τους. Μία από τις τελευταίες εξελίξεις είναι ο διορισμός του νέου πρέσβη, του κυρίου Μπούριαν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον διόλογο με τις περιφερειακές οργανώσεις και με, για τις σχέσεις ε, με ε, διεθνείς οργανισμούς ε, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Στους τομείς της παιδείας, του κράτους δικαίου, του περιβάλλοντος και των υδάτων έγιναν αναφορές σήμερα. Υπάρχει μια κοινή βούληση των χωρών αυτών να εντατικοποιηθούν οι δυνατότητες ε, εργασίας των, ε, των εμπλεκομένων εμπειρογνωμόνων στις διάφορες μορφές περιφερειακής συνεργασίας. Έγινε στη Ρήγα στις 21 Ιουνίου συνάντηση υπευθύνων της Κεντρικής Αθίας ε, για την εκπαίδευση και στο Μιλάνο αντίστοιχα τον Οκτώβριο για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων ε, απαιτείται να υπάρξει ένα σαφές επενδυτικό ελκυστικό κλίμα, καταπολέμηση της διαφθοράς, σταθερότητα των νομικών διαδικασιών, όλα αυτά έχουν σημασία και θα συγκεντρώσουν την προσοχή μας. Τέλος, δίδεται προτεραιότητα στην περιφερειακή σταθερότητα και την περιφερειακή συνεργασία ε, το φόρουμ το οποίο έχουμε θα είναι ένα θα έλεγα ικανοποιητικό φόρουμ έτσι ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος και το 16. Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους πρωτοβουλίες στον τομέα του κράτους δικαίου. Υπάρχουν δύο προγράμματα τα οποία ελπίζουμε ότι είναι αποτελεσματικά. και έτσι θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στην περιοχή αυτή και με τις περιφερειακές οργανώσεις. Από την ΤΕΦΚΟ τώρα ο κύριος Χες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αρχή της διαφοροποίησης είναι σημαντική για τη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές για το Καζακστάν δεν δίνουμε πλέον διμερή βοήθεια, απλά ωφελείται από περιφερειακά και θεματολογικά προγράμματα. Για το Τουρκμενιστάν υπάρχει μια πίστοση 37 εκατομμυρίων ευρώ η οποία θα σβήσει το 18 γιατί είναι και αυτή σχετικά χώρα υψηλού επίπεδου. Παρενέβημεν μεν σε τομείς επαγγελματικής κατάρτισης και σε άλλες χώρες αντίστοιχα έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν ε, θέσεις απασχόλησης και να ξεπεράσουν ε, την έλλειψη δυνατοτήτων λόγω ναι. της ένδυας. Έχουμε διμερεί προγράμματα για τις χώρες αυτές, αναφέρθηκε το τι κάνουμε με αυτές. Έχουμε και κάποια περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα σε άλλους κεντρικούς τομείς όπως το περιβάλλον, το κράτος δικαίου κτλ θα πρέπει να το δούμε αυτό συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα. Έχουμε περιορισμένα μέσα στη διάθεσή μας. Συνολικά έχουμε κάτι παραπάνω από ένα δις. Ε, έχει αυξηθεί κατά 56% τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα πρέπει να στοχεύσουμε καλύτερα στις χώρες αυτές να δούμε πού υπάρχουν ανάγκες και πώς θα τονώσουμε την αίσθηση της ιδιοκτησίας των προγραμμάτων. Έχουμε επαφές στενές με την κοινωνία των πολιτών. Κάποιες κυβερνήσεις από τις χώρες αυτές δεν είναι ικανοποιημένες ε, για αυτές τις επαφές, αλλά θα συνεχίσουμε να τις έχουμε. Αναφέρθηκαν επίσης ε, επί ότι έγιναν βήματα προόδου στον τομέα καταπολέμησης ασθενειών όπως η θυματίωση. Ε, η συνάδελφος αναφέρθηκε ε, σε συγκεκριμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων ε, και γενικά έχουμε συγκροτημένα προγράμματα στον τομέα της υγείας. Ακριβώς επειδή είναι πολλά τα θέματα προσπαθούμε να έχουμε ένα στρατηγικό διάλογο, μια συγκεκριμένη εν περιπτώσει λογική βοήθεια και σε επίπεδο προϋπολογισμού έτσι ώστε να υπάρξει σύνολη βελτίωση του συστήματος. Αυτό δεν θα γίνει εύκολα, θα απαιτήσει χρόνο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή κατανοώντας ότι η αλλαγή στον τομέα αυτό επέρχεται μόνο με πάρα πολύ αργή ταχύτητα. Όπως είπαν πολλοί από τους συναδέλφους σας, δεν μπορούμε εμείς να αυξήσουμε το στρατηγικό διάλογο αλλά τη μόχλευση για μεταρρυθμίσεις όπως στον τομέα της υγείας. Αναφερθήκατε στο θέμα της παιδικής εργασίας και της δουλείας στο Ουσμπεκιστάν. Μειώνεται το πρόβλημα από ό,τι μαθαίνουμε για, την, για τα παιδιά, αλλά το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας είναι σοβαρό θέμα εμείς εγκρίνουμε στην παρούσα φάση ένα πρόγραμμα για την παρακολούθηση της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουσμπεκιστάν. Ε, και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια. Έχουμε ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Παγκόσμια Τράπεζα και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτά. Okay, thank you very much and for clarifying some of the issues, both of you, um, to colleagues. to um, give the floor back. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή και πάλι. Αλλά πάντως να σας ενημερώσω ότι όλες οι μεταφράσεις έχουν ετοιμαστεί σε όλες τις γλώσσες. Είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που το μαθαίνω ότι οι μεταφράσει είναι όλε έτοιμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτέ τι πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις και προτάσεις που έκαναν. Ε, όπως θα θυμάστε, πρόκειται για γνωμοδότηση. Ε, γνωμοδότηση, επομένως, είναι περιορισμένο ο χώρο που έχω στη διάθεσή μου. Ε, εγώ μακάρι να μπορούσα να συμπεριλάβω και περισσότερα. Δύο-τρία πράγματα θέλω να αναφέρω. Οι περισσότεροι συνάδελφοι νομίζω ξέχασαν την σημασία που έχει η Ρωσία, γιατί εμά, ε, όποιο και είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες αυτές, η παρουσία της στην περιοχή θα θεωρηθεί από τη Μόσχα σαν πρόκληση. Επομένως, όσο καλύτερη συνεργασία έχουμε με τη Μόσχα, τόσο το καλύτερο. Δεν θα είναι εύκολο φυσικά, αλλά πάντως είναι και προς το συμφέρον μας. Ή, εν πάση περιπτώσει, ε, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε σχέδιο έχουμε εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτόν τον παράγοντα. Για το ζήτημα τώρα της διαφθοράς. Αυτό συνδέεται έντονα με τη δομή την κοινωνική που βασίζεται στην ε, οικογένεια, στην ευρεία οικογένεια και είναι μια κοινωνική δομή που εμά μπορεί να μας ξενίζει αλλά είναι αυτή που ακολουθείται στις περιοχές αυτές και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ε, υπάρχουν διαφορετήσεις μεταξύ των κρατών, στο... μεταξύ του και ε, για παράδειγμα. Επομένως το ζήτημα είναι και πολιτικό και οικονομικό. Υπάρχουν χρήματα, αλλά αυτά απλώς ε, χρησιμοποιούνται για να ε, διονύζεται ε, η δύναμη ορισμένων οικογενειών. Ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός έχει χρησιμοποιηθεί ε, ως εργαλείο για να προκληθούν πολιτικές αλλαγές. Υπάρχει και μια επιρροή από τις γειτονικέ ε, χώρες, από το Αφγανιστάν κυρίως. Ε, πληθυσμοί από το Αφγανιστάν και αποκορισμένες από τις χώρες εκείνες μιλούν και εκείνες γλώσσες ή γλώσσες που μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλον. Συμφωνώ με τους συναδελφούς οι οποίοι τονίζουν το ζήτημα της υγείας και της περιθάλψης. Ε, γνώριζε για την Ελληνοσία, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζε για το ζήτημα της φυματίωσης στις περιοχές αυτές. Το ζήτημα επίσης είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το εμπόριο διεθνώ ε, δεν ευνοεί τις περιοχές εκείνες της Κεντρικής Ασίας. Το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε και αν λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό ίσως έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συνήθως οικογενειακές. Αναφερθήκατε στη σημαντική της διαφοροποίησης και πράγματι συμφωνώ. Επομένως, σε περιφερειακό επίπεδο θα έπρεπε να επιλύονται και οι, ενδο... Ε, εσωτερικές σε αυτήν την περιφέρεια συγκρούσεις. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 11 η ώρα αύριο το πρωί, ενημερώνει η Πρόεδρος. Και ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα, την αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα, που βεβαίως συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο συγητής μας είναι ο κύριος Σεβαστιά. Έχετε το λόγο. Buenos días, muchísimas gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να πω ότι αυτή είναι η πρώτη γνωμοδότηση για την οποία είμαι υπεύθυνος Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να τους ζητήσω όμως και μια κάποια επίκαια. Έχουμε δύο θα έλεγα συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς η βιοπικιλότητα είναι ζωτική θα έλεγα για πάρα πολλούς ανθρώπους, για πάρα πολλούς ε, για πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους αγρότες στις ε, υποανάπτυξες χώρες, στις φτωχές χώρες, στις χώρες του Νότου. Ε, η βιοπικιλότητα βοηθά να αποφευχθεί η φτώχεια. Είναι μια βασική δραστηριότητα που αποτρέπει από την υπερσυγκέντρωση των πληθυσμών στις αστικές περιοχές και ε, βοηθά πολύ να ξεπεραστούν κάποια από τα προβλήματα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για την καταναλωτική μας συμπεριφορά εδώ και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές με τη συμπεριφορά μας. Καταρχάς η χρήση της βιομάζας ε, σαν ε, καύσιμο, σαν βιοκαύσιμο ε, και επίσης θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μακροπρογράμματα, σε εισαγωγικά προγράμματα μακράς προοπτικής ε, για την λεγόμενη αγροτοβιομηχανική παραγωγή. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, χρησιμοποιώντας ε, και τις δυνατότητες που έχουμε στα πλαίσια των ε, προτύπων κατανάλωσής μας. Δεν θα πρέπει οι προτάσεις μας οι εμπορικές να είναι απειλή για τις χώρες αυτές σε σχέση με τα θέματα βιοπικιλότητας. Υπάρχει το θέμα του ελέγχου της χρήσης της σποράς των παραδοσιακών τρόπων χρήσης της σποράς από πλευράς των γεωργών ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να τις ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν τα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει λοιπόν επίσης και το θέμα της απελευθέρωσης των εμπορικών σχέσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς που λειτουργεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια. Ε, ε, οι διαφορετικές απόψεις δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο ε, χώρο εδώ διακίνησης παρόλα αυτά θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα συμπληρώσουν το κείμενο είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει την βοήθεια σε δραστηριότητες αρνητικές για τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων της στον τομέα της ε, παραγωγής ενέργειας, στον τομέα της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας επίσης και στα πλαίσια της αντιμετώπισης ε, των προβλημάτων που δημιουργούν οι κλιματολογικές αλλαγές θα πρέπει να μεταφέρει τις απόψεις αυτές και στις υπόλοιπες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε έτσι ώστε να προκαλέσουμε κάποιες θετικές αλλαγές στην πολιτική συνεργασία και ανάπτυξης που έχουμε με τις χώρες αυτές. Είναι ένα θέμα πολύ θα έλεγα ενδιαφέρον, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί σε βάθος αλλά η βιοπικιλότητα πρέπει να διατηρηθεί γιατί επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι σχέσεις μας οι οικονομικές μαζί τους είναι ιδιαίτερα εύθραστες και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σύντομα. Ελπίζω λοιπόν ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, θα είναι θετική για τις ε, κατευθύνσεις της γενικότερης της πολιτικής μας. Ε, σίγουρα είναι η πρώτη σας νομοδότηση, αλλά είναι σαφές ότι γνωρίζετε όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Λοιπόν, ο κύριος Γκουερέρο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να καλωσορίσω τον κύριο Σεμπαστιά, ο οποίος έχει την ίδια αν θέλετε επαγγελματική προέλευση με μένα στην Ισπανία και σίγουρα είναι σαφές ότι υπάρχει μια επίοικια απέναντι σε αυτούς που για πρώτη φορά καταθέτουν μία πρόταση είτε εδώ είτε στην Ολομέλεια. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από αυτή την φιλική στάση, να μην περιοριστούμε σε αυτό, αλλά όπως είπε και η Πρόεδρος, τίθεται το θέμα της βιοπικιλότητας, διότι επηρεάζει τους πάντες επηρεάζει τους πάντες ε, με πολύ έντονο τρόπο, με πολύ κρίσιμο τρόπο και επηρεάζει σε καθημερινή βάση όλες τις προσωπικές εμπειρίες σε γεωγραφικά επίπεδα διαφορετικά που οδηγούν μερικές φορές σε καταστροφές στον τομέα της βιοπικιλότητας, συνέπειες των ενεργειακών πολιτικών, των κλιματολογικών αλλαγών, των εμπορικών δραστηριοτήτων και όπως ε, είπαμε ο κύριος Σεμπαστιά που δεν είναι αν θέλετε ιδιαίτερα τακτικό μέλος αυτής της Επιτροπής φαίνεται όμως ότι αναγνωρίζει ότι εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της συνέπειας της αναπτυξιακής, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να είναι εγκάρσια συνεκτική και με την πολιτική των εμπορικών σχέσεων και με την πολιτική του περιβάλλοντος και με θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα, ευάλωτα Γι' αυτό λοιπόν Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία που έχει το θέμα αυτό στην εξέλιξη της σημερινής κοινωνίας, ένα θέμα το οποίο επίσης και πολιτικά έχει μεγάλη σημασία για ό,τι απασχολεί την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Μελετήσαμε με μεγάλη προσοχή το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ένα πρόβλημα που βρήκα για τα κριτήρια βιωσιμότητας της ε, βιομάζας της ε, περιφέρειες της Ευρώπης. Πιστεύω πως στην έκθεσή μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς θα βελτιώσουμε την βιωσιμότητα της δασοπονίας Στον τομέα αυτό, στη χώρα μας, έχουμε μια πολύ καλή βιώσιμη πολιτική, πολιτική βιωσιμότητας. Έχουμε κριτήρια βιωσιμότητας και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης είναι και θέμα και επικουρικότητας. Στη Φιλανδία έχουμε διαφορετική δασική πολιτική και η συνοχή φυσικά παίζει και αυτή ένα ρόλο, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Θα ήθελα λοιπόν να διαγραφεί αυτή η εσωτερική άποψη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης από την έκθεση και να επικεντρωθούμε στην αναπτυξιακή πολιτική προώθησης της ε, βιωσιμότητας και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έπειτα υπάρχει και κάτι που είναι πάρα πολύ αντιφατικό και εμείς θα υποβάλουμε τις δικές μας ε, τροπολογίες και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα αντιφατικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, συμφωνώ κι εγώ με τα σημεία 4 και 5 συγκεκριμένα που αναφέρονται στα ουδέτερα κριτηρία βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα. Εργάστηκα κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία για αυτό θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χθε είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ για την αναπτυξιακή ε, πολιτική συνοχής και είναι κάτι που πολλές φορές παραμελούμε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ε, βιοκαυσίμων. Πολλές φορές έχουμε καλές προθέσεις, αλλά αυτές οι καλές προθέσεις δημιούργησαν προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό με απασχολούν πάρα πολύ αυτά τα θέματα, το θέμα της βιομάζας ε, στην ε, δασοπονία. Βέβαια έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούμε να του ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα δώσω τώρα το λόγο την Ρέκε Χάουζερ από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις προτάσεις που ακούσαμε και τον ευχαριστώ και για την προσοχή που έδωσε στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, στρατηγικής βιοποικιλότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βιοπικιλότητα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μας θα λάβουμε τα σχόλιά σας. Τώρα, κριτήρια βιωσιμότητας για την δασοπονία. Δυστυχώς θα πρέπει να επανέλθω και να απαντήσω στον εισηγητή αργότερα, διότι δεν είναι ένα θέμα των άμεσων αρμοδιοτήτων μου αυτή τη στιγμή. Και από, από όσο ξέρω αυτό το θέμα υπάγεται στην ε, οδηγία για τις ε, ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, για τα βιοκαύσιμα. Γι' αυτό λοιπόν θα επανέλθω και θα σας ενημερώσω για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργασίες μας. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Έχουμε τον κύριο Ζακ Τισμούτ από την ΓΑΜΑΒΕΛΤΑ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου αυτή την έκθεση και το προσχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναπτυξής. Όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση δασών, Εδώ θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι εδώ και μία δεκαετία η στρατηγική επιλογή της Κομισιόν ήταν να ε, στοχεύσει κυρίω στο ζήτημα της διαχείρισης των δασών μέσω της FLECT, το οποίο δεν ε, συνδέεται άμεσα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την βιώσιμη διαχείριση, αλλά συνδέεται και δημιουργήσαμε εταιρικέ σχέσεις με χώρες αναπτυσσόμενες που το επιθυμούσαν, έτσι ώστε να εξηγιανθεί ο τομέας της δασοπονίας, να βελτιωθεί η χνελασιμότητα από την παραγωγή της ξυλίας μέχρι το τελικό προϊόν και να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία υφίσταται και συμπεριλαμβάνει και υποχρεώσεις ε, βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησε να προωθήσει τον στόχο της βιωσιμότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τώρα. Συμμερίζομαι όμως τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ότι πράγματι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε. Κύριε Σεβαστία, αν θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις σας. Φυσικά θα συμπέσουμε στα θέματα αυτά τα οποία αναφέρε ο κύριος Γκουερέρο Σαλόμ. Υπάρχει το θέμα του εύθραυστου χαρακτήρα ή του ευάλωτου χαρακτήρα των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε εξαιρετικά ευάλωτες καταστάσεις τίθεται το θέμα της άμεσης αναφοράς στο θέμα της βιομάσας, θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και ξεκάθαροι λέγοντας ότι η υποστήριξη στην κατανάλωση της βιομάζας είναι κάτι το οποίο στην ουσία πρέπει να σημειωθεί ότι λειτουργεί αρνητικά ε, για την προστασία της βιοπικιλότητας. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αλλάξουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως είναι σαφές ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μία συνένεση εδώ και σε σχέση με τη βιομάζα και ε, με τα βιοκαύσιμα είναι δύο θέματα τα οποία συνεισφέρουν αρνητικά ε, στο θέμα της προστασίας της βιομάζας θα προσπαθήσουμε λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την διατύπωση μιας έκθεσης ε, σαφούς και αποδεκτής από όλους. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών αύριο στις 10. Τελειώνουμε για σήμερα, ξεκινάμε με ψηφοφορίες στις 3. Η έκθεση Γκουερέρο θα είναι η τελευταία ε, στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις. Καλή τύχη.